Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής ως συνήθως. Να σας προειδοποιήσω ότι αναμεταδίδεται η συνεδρίασή μας από το διαδίκτυο. Δύο θέματα έχουμε. Το πρώτο αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού 966 του 12 σχετικά με την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Θέτουμε πρώτα σε ψηφοφορία την τροπολογία 12. Ποιοι είναι κατά αποχές δεκτή. Η επόμενη τροπολογία, η 13, έχει αποσυρθεί. Δεν θα ψηφιστεί συνεπώς. Και μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα την 14 Σόλτς. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ακολουθεί η συμβιβαστική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συνεχίζουμε. Περνάμε στην 2 γιατί όπως είπα οι 15 και οι 16 έχουν ήδη καλυφθεί. Οι 2 τώρα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τρία. ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ventuno. Sì. 21 è identica al 22, quindi praticamente vale. Λοιπόν, υπέρ της 22, κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8. Έχει ζητηθεί ε, κατά ψηφοφορία εδώ. Το πρώτο τμήμα χωρίς να τεθεί το θέμα του 22-7 και το δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και τώρα η υπόλοιπη φράση, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 24 καλύπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 26 Σόλτς υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα για μια στιγμή στην εννέα. στην εννέα. ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το υπολογία δέκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές 15 υπέ, 5 κατά, κανένας αποχή. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον συνάδελφο. Η άλλη ψηφοφορία αφορά θέμα για το οποίο είμαι εγώ εισηγητής. Η Επιτροπή Ανάπτυξης, όπως ξέρετε, ζήτησε από την Επιτροπή μας να κάνει μια ερμηνεία του κανονισμού για να διευκρινιστεί αν οι γενικοί κανόνες οι οποίοι έχουν καθοριστεί για τη σειρά των τροπολογιών στην Ολομέλεια, άρθρα 156 και 161, πρέπει να εφαρμόζονται και στις ψηφοφορίες στις κοινοβουλευτικές επιτροπές σχετικά με τις προφορικές τροπολογίες. Τρεις ερωτήσεις. Μπορεί κανείς να τροποποιήσει άλλη τροπολογία με προφορική. Η δεύτερη ερώτηση. Είναι πάντα υποχρεωτικό να τίθενται σε ψηφοφορία οι προφορικές ακόμα και αν δεν υπάρχει ε, κάποιος που είναι κατά ή θεωρούνται αυτόματα έτσι δεκτές. Και τρίτον, ποια είναι η σειρά, ποια είναι η τάξη αν θέλετε που ακολουθείτε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Εσείς έχετε ε, το έγγραφο μπροστά. Το άρθρο 156 δεν προβλέπει τροπολογήσεις των τροπολογιών. Το προφορικό η προφορική τροπολογία αφορά την τροπολόγηση του κειμένου και αντικαθιστά ένα τμήμα του κειμένου, δεν αλλάζει όμως την ουσία. Στην περίπτωση τώρα που τεθεί προφορικά μια νέα τροπολογία ή ε, να προταθεί μια διόρθωση μιας άλλης τροπολογίας, το θέμα και στις δύο περιπτώσεις αφορά την τροπολόγηση του κειμένου. Τώρα, για το επίπεδο και τη στάση της αντιπολίτευσης. Η πρακτική είναι 40 ε, θα έλεγα βουλευτές. Δεν μπορεί να γίνει δεκτή αν 40 βουλευτές είναι κατά, δηλαδή μιλάμε περίπου για το 5%. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε αν οι προφορικές τροπολογίες, ακόμα και οι μη μεταφρασμένες συμβιβαστικές τροπολογίες, μπορούν να απορριφθούν αν το 1 πέμπτο των μελών είναι κατά. Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψή μου. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να απαντήσουμε όπως σας το έχω περιγράψει. Τώρα, στην περίπτωση που δεν απορριφθεί μια προφορική τροπολογία, το αν θα πρέπει δεν θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία ή να θεωρηθεί αυτόματα ότι έχει γίνει δεκτό, δεν αλλάζει τίποτα. πρέπει να ψηφιστεί ίσως και δεν θα πρέπει ο πρόεδρος να αποφασίζει κάθε φορά. Και σε αυτό το θέμα η γνώμη μου είναι αυτή και θα πρέπει να συνενέσετε εφόσον βέβαια το θέλετε. Ο κύριος Ντάφ έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι σαφές πως ε, διαφορετικές επιτροπές ε, το προσεγγίζουν διαφορετικά. Νομίζω πως ο κανόνας του 5% για την Ολομέλεια πρέπει να ισχύσει και στην Επιτροπή για να έχει κανείς αντίρρηση σε μια τροπολογία ή προφορική τροπολογία. Αλλά πρέπει νομίζω να οριστεί αυτό ρητός, όχι να είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Πρόεδρου της Επιτροπής και επίσης θα ρωτούσα, χωρίς να έχω κάποια απάντηση, το εάν θα δοθεί στον εισηγητή ένας ιδιαίτερος ρόλος στο να καθορίσει το εάν θα δεχτεί όχι τις προφορικές ε, τροπολογίες ε, επί των τροπολογιών. Σε, περίπλοκους, σε περίπλοκα θέματα υποθέτω ότι ο συγητής μπορεί να κρίνει το εάν ε, θα επιτρέψει ε, προφορική τροπολογία επί τροπολογίας οπωσδήποτε ο εισηγητής πρέπει ε, να ερωτηθεί οπωσδήποτε για την άποψή του επί του θέματος πριν ε, αποφασίσει η Επιτροπή. Προτείνω να τα γράψουμε αυτά στην επιστολή ότι κανονικά ο συγητής ε, πρέπει να ρωτάτε Επομένως, στην ουσία κύριε Ντάφ, ζητάτε διόρθωση ε, της επιστολής που νομίζω ότι σας έχει διενεμηθεί. Εντάξει, τώρα το ότι θα πρέπει να είναι μέλος της Επιτροπής ε, αυτός ο οποίος ενδεχομένως θα αντιταχθεί, ναι, όπως και οποιοδήποτε άλλο μέλος της Επιτροπής, αλλά εάν η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει εκ των υστέρων, ε, αυτό είναι αυτονόητο. Είναι σωστή η παρατηρήσή σας, αλλά νομίζω ότι ήδη περιέχεται στην γραπτή απάντηση την οποία προετοιμάσαμε παρόλα αυτά. Εάν θεωρείτε ε, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί ρητά, ε, τότε ναι, μπορούμε να το γράψουμε ρητά και κατηγορηματικά και ε, να μην ψηφίσουμε σήμερα. Εάν έτσι αποφασίζετε και αν ε, εάν όμως όλοι πιστεύουν και ο ίδιος ο κύριος Ντάφ ότι θεωρείται αυτονόητο ε, αυτό που λέει, να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία των ψηφοφοριών και μπορούμε να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Προέδρου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 scritto vuol dire non si fa parere, non si fa parere. Mm-hmm. Qui, qui, questi sono tutti chiamati Allora, Λοιπόν, συνεχίζουμε τις εργασίες της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα ανακοινώνω επίσημα στην Επιτροπή αυτά που ήδη γνωρίζετε όλοι φαντάζομαι, γιατί οι περισσότεροι μεταξύ μόνοι είστε παρόντες στους συντονιστές. Παρ' όλα αυτά σας λέω ότι όσον αφορά το αίτημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης δύο ε, κομμάτων ε, με τις αξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίστηκε να ξεκινήσει, να ληφθεί η απόφαση για την άναξη των διαδικασιών στην επόμενη συνεδρίαση έτσι ώστε να έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και το υλικό που είναι απαραίτητο έτσι ώστε να ληφθεί σωστά η απόφαση. Επί του σημείου 2, ε, διαρθρωμένος ε, διάλογος το σημείο 2 της συνέδριας των συντονιστών, αποφασίσαμε να αποστείλουμε επιστολή στον Επίτροπο Σεύκοβιτς, ο οποίος ε, είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος να συμμετάσχει στις συνεδρίες του Μαΐου, έτσι ώστε ε, να ε, μας δηλώσει αν έχει διαθεσιμότητα για κάποια άλλη συνεδρία της Επιτροπής, να παραστείλει σε κάποια άλλη συνεδρία της Επιτροπής. Η Επιτροπή ε, έδωσε την ε, αρμοδιότητα στον Πρόεδρο να υποβάλει προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 59 και σε συνεργασία με την Λίμπε και τη Γιούρη όσον αφορά την υλοποίηση ε, του προγράμματος της Στοκχόλμης επί του οποίου είχαμε κάνει κοινή έκθεση έτσι ώστε να μάθουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία, ποιες είναι οι δυσκολίες που ενδεχομένως έχει συναντήσει η διαδικασία. Θα πρέπει να γίνει άμεσα η γνωμοδότηση αυτή, αλλά ε, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον ε, μήνα Μάιο. Ε, όμως να θυμίσουμε ότι ήδη βάσει του άρθρου 51 έχει δοθεί αρμοδιότητα στις τρεις επιτροπές από κοινού να εκπονήσουν έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα του Στοκόλμης και την ενδιάμεση αναθεώρηση. Επίσης ε, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή δεν θα εκφράσει γνωμοδότηση επί των τροποποιήσεων της ε, δημοσιονομικής ε, πειθαρχίας, γιατί δεν υπάρχουν θέματα θεσμική, θεσμικού ενδιαφέροντος. Όμως, όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων, το ΕΛΚΕ θα αναλάβει την έκθεση. Ο Αντιθέτως, ο εισηγητής γνωμοδότησης ε, όσον αφορά την καλύτερη νομοθέτηση νομίζω ότι Α, ε, νομίζω ότι είναι αρμόδια ε, η Επιτροπή Προϋπολογισμού, όχι η ΛΥΜΠΕ, και θα είναι εισηγητής από την ομάδα FD. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω στις ανακοινώσεις και επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε με την εξέταση του ε, ε θέματος 11 δηλαδή δημοσιονομικές επιπτώσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων. Εδώ θέλουμε γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και η επί της ουσίας είναι ο συνάδελφος Έλλης η έγκριση της Επιτροπής Προϋπολογισμών προβλέπεται τον μήνα Ιούλιο. Επομένως, μέχρι τις 28 Μαΐου εμείς θα πρέπει να έχουμε εκπονήσει τη γνωμοδότησή μας. Το σημείο έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης. Αλλά δεν έχουμε ακόμα τον εισηγητή. Ναι, αλλά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε σήμερα έπρεπε να ξέρουμε τον εισηγητή. Ε, το ΕΛΚ είχε ζητήσει να αναλάβει την έκθεση, αλλά ακόμα δεν έχουμε όνομα, επομένως θα πρέπει να αναβάλουμε την εξέταση του σημείου αυτού. allora. Sì, sì. Ecco, e του σημείου μπορούμε να επιστρέψουμε στην ημερήσια διάταξη την αρχική μας έτσι ώστε να συζητήσουμε το σημείο 6 προϋπολογισμός 2010 εντολή για τον τριμερή διάλογο ε, που η αντικαταστάτριά μου κυρία Λεγκρίπ αποφάσισε από κοινού την Επιτροπή ε, να αναβάλει χθε και να την εξετάσει σήμερα. Προπολογισμό 2014 λοιπόν, εντολή για τον τριμερή διάλογο. Οι επιτροπές, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να δώσουν πρώτα κάποιες γενικές κατευθύνσεις όσον αφορά τον, ε, την εντολή αυτή και μετά μπορούν να παρέμβουν ενδεχομένως μέσω υποβολής τροπολογιών. Μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και με την κυρία Γιάνσεν. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ, ο οποίος ε, θα παρουσιάσει την έκθεση, ε, είναι εδώ. Είναι δύσκολο το όνομά σας, κυρία μου, δεν μπορώ να το προφέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μέσερ Σμιτ, ο οποίος είναι εισηγητής και μετά σε εσάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντιμος μια που το συζητήσαμε το θέμα πριν συνταχθεί η γνωμοδότηση. Σύντομα λοιπόν, ελπίζω να αντικατοπτρίζει τις απόψεις και ιδέες των μελών της Επιτροπής όπως συζητήθηκαν στην συνάντησή μας και ανάμεσα από τα μεταξύ ζητημάτων η συγκεκριμένη γραμμή του προπληγισμού για τις εκλογές, τις ευρωεκλογές του χρόνου, αλλά βεβαίως άλλο ζήτημα αφορά την ε, αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών και την στρατηγική επικοινωνίας στις τελευταίες ε, ευρωεκλογές. Ε, σε αυτό είναι υπερυπολογισμό χρόνου εκλογών, οπότε το βασικό είναι αυτό όσον αφορά την Επιτροπή μας. Οπότε είμαι ανοιχτό στις ε, προτάσεις σας και ελπίζω αν ε, δεν συμφωνούμε πλήρως να μπορέσουμε να εργαστούμε επί κάποιων τροπολογιών και να με υποστηρίξει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, zpráva od Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση Messerschmitt επικεντρώνεται στην λιτότητα, την οικονομία κτλ. Αλλά δεδομένης της κρίσης και του ότι πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη δεν συμφωνώ με τις βασικές ιδέες της έκθεσης. Ο εισηγητής προτείνει την αξιολόγηση των προγραμμάτων όπως το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργών Πολιτών το έτος αυτό πρέπει να προωθήσει την ε, συμμετοχική ιδιότητα των πολιτών σε όλα τα επίπεδα και είναι σημαντικό να έχουμε ε, μόνιμα αποτελέσματα, ειδικά φέτος καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές. Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο των Πολιτών και να γνωρίζουν οι πολίτες ε, τα δικαιώματά τους. Αυτό σημαίνει κονδύλια για επικοινωνία, αλλά φοβάμαι πως η αξιολόγηση της Ευρώπης ε, των πολιτών δεν θα είναι δυνατή δεδομένων των κονδυλίων που έχει διαθέσει το Συμβούλιο. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να τονίσουμε το ότι ο προπολογισμό του 2014 πρέπει να είναι υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αυτό μπορεί να γίνει με την αύξηση των κονδυλίων και αύξηση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματική και πρακτικής κατάρτισης. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη για να εξηγηθούν τα δημόσια οικονομικά. Ένας μειωμένος ευρωπαϊκός προπολογισμός είναι αντίθετος με αυτούς τους στόχους. Επίσης πρέπει να σημειώσω πως στο τέλος του 2012 δεν υπήρχαν πιστώσεις πληρωμών και πρέπει να μεταφερθούν από το 2012 στο 2013 και μιλάμε για πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε πρέπει νομίζω γρήγορα να τροποποιήσουμε τον προτινόμενο προπολογισμό για να μην έχουμε πάλι νέες μεταφορές στο έτος 2014. Τέλος, ήθελα να σχολιάσω το σχέδιο ιδίων πόρων της ε, Κομισιόν, μεταρρύθμιση δηλαδή του ΦΠΑ και νέο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά για την γνωμοδότηση για τον προπολογισμό του 2014 και θα τα συμπεριλάβω στις ε, τροπολογίες μου. Έφνα και στα παρόλα. Ευχαριστώ κύριε Σκέφνερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί νομίζω πως επί της αρχής θα έχουμε συζητήσει τα πράγματα πολλές φορές οπότε δεν θα αναφερθώ σε ζητήματα αρχών θα αναφερθώ μόνο συγκεκριμένη πρόταση του κυρίου Μέσσερ με την οποία συμφωνώ επί της αρχής υπάρχουν κάποια πράγματα δύο βασικά για τα οποία θα να κάπως διαφορετικές ε, διατυπώσεις ε, μπορώ να σας τα πω αμέσως. Έχουμε το σημείο 4 και ευχαριστώ τον εισηγητή για το ότι έβαλε εδώ πέρα την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών και το σχετικό πρόβλημα. Εκεί όπου λέει όμως ε, need for priority in the budget ε, εκεί που λέει ανάγκη για προτεραιότητα όχι μόνο για τις πρωτοβουλίες αλλά και για την επικοινωνία Δεν θα ανέφερα λοιπόν μόνο τις ε, πρωτοβουλίες αλλά όπως είπε και ο συνάρχος Μπρος Μποχάτα ε, νομίζω πως οι ε, συνάρχος νομίζω πως και η ίδια η Κομισιόν με την προσέγγιση της και το προσωπικό δεν μπορεί να παρακολουθήσει ε, σωστά την Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία. Αυτή είναι μια ευκαιρία για όλους τους Ευρωπαίους να αναμειχθούν, να μιλήσουν. Εάν δεν το δούμε και νομικά και τεχνικά καλύτερα στο μέλλον και για όσον αφορά τη διαχείριση της υπηρεσίας αυτής, τότε θα έχουμε μια αποτυχία. Γι' αυτό χρειάζεται όντως περισσότερα λεφτά και θα πρότεινα να συμπληρώσουμε επικοινωνία, διαχείριση και στήριξη από την Κομισιόν. Το άλλο σημείο είναι το σημείο 7 έτσι κάπως πιο γενικό. Και νομίζω πως ε, σωστό είναι να αναφέρομαι πως σε μια εποχή από την οποία απαιτούμε από πάρα πολλά να κάνουν οικονομία, το ίδιο μπορεί να ισχύσει και για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δηλαδή, αν είναι να μην τονίσουμε μόνο τη μία πτυχή αλλά ολόκληρο το σύνολο πρέπει ταυτόχρονα να πούμε πως και θα το πω στα αγγλικά έχω διατυπώσει μια τροπολογία με τις αυξανόμενες ευθύνες και αρμοδιότητες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται τα τα μέσα και ε, τους δικούς του πόρους αλλιώς δεν θα μπορούμε να είμαστε σε θέση πραγματικά να εκπληρώσουμε τη την αποστολή μας. Οπότε εγώ θέλω, θα ήθελα να αναφερθούν και οι δύο πλευρές. Για το πρώτο δε της πρωτοβουλίας των πολιτών είμαι σίγουρος πως κάτι θα κάνει ο εισηγητής. Ε, Αλλιώ ε, τώρα για το δεύτερο δεν ξέρω μπορεί να καταθέσουμε όπως είπα μια τροπολογία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Εφνερ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νταφ. Κύριε Πρόεδρε, στην παράγραφο 3 ο εισηγητής ε, κάνει λόγο για αξιολόγηση της ε, στρατηγικής επικοινωνίας για τις εκλογές του 2009. Νόμιζα πως ε, ήδη είχαμε δει κάτι τέτοιο και είχε υπάρξει σχετική αναφορά. Και μια που έχουμε εκλογέ του χρόνου, και μιλάμε για τον προπολογισμό του 2014, μήπως θα έπρεπε να ζητήσουμε μια αξιολόγηση της ε, στρατηγική επικοινωνία για τις ευρωεκλογέ του 2014. Δεν νομίζω πως υπάρχει ε, κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το εξακριβώσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Μέσσερ Σμιτ, εσείς τώρα θα μας ε, απαντήσετε και θα βγάλετε και τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Και μετά από αυτά που είπε ο πρώτος ομιλητέ, νομίζω ότι αυτά τα οποία υπέχουν σημασία, αλλά δεν ξέρω αν είναι η σωστή θέση η γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ ή θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη έκθεση στο τέλος όταν φτάσουμε στην Ολομέλεια. Για τον κύριο Χέφνερ αναφερθήκατε σε δύο πράγματα. Το πρώτο, σε σχέση με το σημείο 4, μπορούμε να δούμε τι πώς θα προχωρήσουμε. Είχαμε κάποια επιμελητιακά θέματα εδώ στη σύνταξη και ίσως μέσω της τροπολόγησης του κειμένου θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση σχετικά με τους πόρους. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να τεθεί στην τελική έκθεση, στην Ολομέλεια και όχι στην γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις πρωτοβουλίες που έχουμε μπροστά μας. Και τέλος, για ε, τον κύριο Νταφ. Εγώ προσπάθησα να προχωρήσω σε μια αξιολόγηση του τι έγινε ε, το, ε, από το 2009 και το 2009 με τις εκλογές έτσι ώστε να δούμε τι θα έπρεπε να διορθώσουμε και τι να αφήσουμε και να έχουμε μια πλήρη στρατηγική για τις, για τις επόμενες εκλογές και την προεκλογική εκστρατεία. Συμφωνώ λοιπόν με την ιδέα, το θέμα είναι πώς θα το διατυπώσουμε σωστά. Πάντως θα βρεθεί τρόπος, είμαι σίγουρος. Καλώς. Η γνωμοδότηση αυτή θα πρέπει να γίνει δεκτή στις 28 Μαΐου στη συνεδρίασή μας. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών η Τετάρτη 8 Μαΐου 12η μεσημβρινή. Λοιπόν, στα διάφορα φτάσαμε, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Να υπογραμμίσω την επόμενη συνεδρίασή μας, 27 Μαΐου, από τις 3 μέχρι τις 6.30 και 28 Μαΐου από τις 9 μέχρι τις 12.30. Πέρα της συνεδρίασης, θα συνεχίσουν μόνο οι συντονιστές για να κλείσουν τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει.